Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση. Ο πρόεδρος Ζαν Κλοντ Γιούγκερ χθες μας ενημέρωσε για τη σύνθεση της Νέας Επιτροπής και την ε, κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Επιτρόπων. Η διάσκεψη των Προέδρων των ε, Επιτροπών συνήλθε χθες το βράδυ και καθόρισε μια πρόταση απόφασης η οποία θα υποβληθεί στην διάσκεψη των Προέδρων των ομάδων, των πολιτικών ομάδων σήμερα, για τις ειδικέ αρμόδιες επιτροπές για την κάθε ακρόαση των υποψηφίων επιτρόπων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των ακροάσεων αυτών. Η Επιτροπή Προπολογισμών θα είναι αρμόδια για τη διοργάνωση της ακρόασης της κυρίας Γεωργίευα υποψηφίας επιτρόπου για τους προπολογισμούς σε συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου. Ως προς το χρονοδιάγραμμα των ακροάσεων θα λάβουν χώρα στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου καθώς και την 1η Οκτωβρίου και μετά 6, 7 και 8 Οκτωβρίου. Θα ήθελα σε όλες τις συνεδριάσεις που θα συμμετάσχει η Επιτροπή Προπολογισμών να μην συμπέσει με την ψηφοφορία μας για τον προπολογισμό του 2015. επίση, εξέφρασα γραπτός το ενδιαφέρον μας να λάβουμε μέρος στην ακρόαση του κ. Κάιτανεν λόγω των ε, αρμοδιοτήτων που θα αναλάβει σε θέματα προπολογισμού. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που ήθελα να σας κάνω. Τώρα για την ημερήσια διάταξη. Ελπίζω ότι την εγκρίνουμε όλοι. Και εν ώψη της θα δούμε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση τις σχετικές εκθέσεις που αποβλήθηκαν τις περασμένες εβδομάδες. Le premier, le premier rapport qui vient en discussion. Η πρώτη έκθεση που θα συζητήσουμε είναι η έκθεση του κυρίου Εστέμπαν Κοσάλε Πόν, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση στην περιοχή τη Καστίγια Ιλεών στην Ισπανία. Με 700.000 ευρώ κινητοποίηση. Έχετε λάβει τις τροπολογίες. Τροπολογία υπαριθμών 6 καλύπτεται. Δεν θα χρειαστεί να την ψηφίσουμε. Τροπολογία 7 Ο εισηγητής προτείνει να απορριφθεί. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. 13 υπέρ. 15 κατά. Απορρίπτεται. 8. Τροπολογία 8. Καλύπτεται. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. 9. Ο εισηγητή μα προτείνει να απορριφθεί. Υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε. Υπέρ και πάλι. Με συγχωρείτε. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. 15 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται. 10. Καλύπτεται, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Το ίδιο 11, 12 και για το 12. Την πρώτη, δεύτερη, τρίτη τροπολογία. Τροπολογία 4. Ο εισηγητής μας προτείνει να απορριφθεί. Υπέρ, προτείνω να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Όσοι είναι υπέρ, θα πατήσετε το πράσινο κουμπί, το κόκκινο όσοι απορρίπτεται και το λευκό όσοι απέχετε. Τροπολογία 4. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται με 15 ψήφου υπέρ, 13 μάλλον υπέρ, 15. Με συγχωρείτε, ε, λάθος. 15 είναι ψήφοι υπέρ, 13 15 είναι ψηφί κατά, 13 υπέρ και 2 αποχές. Τροπολογία 5. Καλύπτεται, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. Οπότε ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν ανάπαντες. Κύριε Δεβρέ. Με συγχωρείτε πρόεδρε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Η κάρτα μου φαίνεται να μην λειτουργεί. Παρόλο που την έχω. Εψήφισα υπέρ. Πέρας της ψηφοφορίας. 28 ψήφοι υπέρ, στις οποίες θα προσθέσουμε την ψήφο του κ. Διπρέ. 29, 4 κατά, δεν υπάρχουν αποχές. Να δώσω τώρα το λόγο. Όχι, με συγχωρείτε, θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες στο σχέδιο έκθεση του κ. Πολτάρη για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Τροπολογία 6. Δεν θα ψηφιστεί. Τροπολογία 7. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Να ρωτήσω λοιπόν ποιοι είναι υπέρ. Ηλεκτρονικός Ωραία. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Pardon Bon, c'est pas... À Ας ψηφίσουμε λοιπόν ε, διανάταση της χειρός. Υπέρ. Όλοι είναι υπέρ. Κατά. Δεν υπάρχουν ψήφοι κατά. Α, ούτε εποχέ. Εγκρίνεται. 8 καλύπτεται. 9 καλύπτεται. Τροπολογία 10. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. 11. Υπέρ. 12. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. το ίδιο. 13. Ποιοι είναι υπέρ. Δεν υπάρχουν ψήφοι κατά. Α, με συγχωρείτε. Είναι τρεις οι ψήφοι, οι αρνητικές. 14 υπέρ. Ο συγκεκριτής είναι υπέρ, ευχαριστώ. Κατά. 5 ψήφοι κατά. Τροπολογία πρώτη καλύπτεται, δεν θα ψηφιστεί. Δύο. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 3. Καλύπτεται. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Τροπολογία 5. Καλύπτεται. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση με 28 ψήφους υπέρ, 3 κατά και καμία αποχή. 29 με τον κύριο Ντεπρέ. Ας περάσουμε τώρα στην έκθεση τη Λιάντιν Ριάντα, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, τεχνική βοήθεια με 330.000 ευρώ κινητοποίηση. 10, τροπολογία 10, η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο εποχές. Εγκρίνεται. 11. Η εισηγήτρια προτείνει να απορριφθεί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δώδεκα. Η συγκέντρια και πάλι είναι κατά τη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ η συγκέντρια Υπέρ. Ίσως θα μας ε, βοηθήσει εδώ η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 13. Εψήφισαν απαντές. Ο κ. πρέπει κατά. Το σημειώνουμε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ και 6 κατά. 14. Υπέρ η εισηγήτρια. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Τροπολογία 16. Η εισηγητρία είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 17. Είσαι και 31 κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 η είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές, εγκρίνεται. 19. Η εισηγήτρια είναι κατά. Υπέρ. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, θα είναι σαφέστερο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Ο κύριος Δεπρέ είναι υπέρ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η τροπολογία με 17 ψήφους υπέρ και 15 κατά. Τροπολογία 20. Ο εισηγη... Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία πρώτη. Η συγκέντρια, με συγχωρείτε. Τροπολογία πρώτη. Η συγκέντρια υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τρεις αρνητικές ψήφοι. Ποιοι απέχουν. Τρεις αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Η συγκεκριμένη είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχέ. Η τροπολογία εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Είσαι και τρέν υπέρ. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Τρει αποχές. Η τροπολογία 3 εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Είσαι και είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Τροπολογία 5 η συγκεντρίνα και πάλι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ποιοι είναι κατά της τροπολογίας. Αποχές. Δεν υπάρχουν εποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τρει αρνητικέ ψήφοι. εποχέ. Δύο εποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Η τροπολογία 7. Η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά. Αποχές. Τρεις αποχές. Τροπολογία 8. Η συγκεντρία είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Τρεις αρνητικές ψήφοι. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. 9. Η συγκέντρια είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Τρεις αρνητικές ψήφοι. Αποχές. Δύο αποχές. Τρεις αποχές. Για το σύνολο του κειμένου στροποποιήθηκε η Ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. ψήφισαν άπαντε πέρα της ψηφοφορία. Ο κ. Ντεπρέ είναι υπέρ. 26 ψήφοι υπέρ. 3 ψήφοι. Κατά καμία αποχή. Και τώρα θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες του σχεδίου έκθεσης του κυρίου Κίρτσου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. για τις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και την Αττική 6 εκατομμύρια 860.000 ευρώ. Τροπολογία 6 καλύπτεται. 7 όσοι γιατί είναι κατά. Υπέρ. Βλέπω να υπάρχει μικρή διαφορά, οπότε θα έλεγα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. να άπαντες πέρας. Κύριε Ντεπρέ, λειτουργεί τώρα. Ωραία. 17 ψήφοι υπέρ, 15 κατά. Εγκρίνεται. 8. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Η ηλεκτρική ψηφοφορία, όχι δεν χρειάζεται. Ένα δεύτερο χειρός. Ε, υπέρ. Κατά. Δεν υπάρχουν αρνητικέ ψήφοι υπέρ. Ε, αποχέ, συγγνώμη. Ε, δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται. 9. Καλύπτεται. 10 το ίδιο. 11 το ίδιο. 12. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Πιστροπολογία 12. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ε, να απαντήσω. πέρας. Η τροπολογία εγκρίνεται με 17 ψήφους υπέρ και 15 κατά. 13. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αρνητικές ψήφοι. Τρεις αρνητικέ ψήφοι. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται. Ήταν η τροπολογία 13. 14. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Επίσης, ανάπαντες πέρας. Η τροπολογία απορρίπτεται με 20 προς 10 ψήφους. 15. Καλύπτεται. Δεν θα ψηφιστεί. Και η πρώτη τροπολογία. Και η δεύτερη. Το ίδιο και η τρίτη. Στην τροπολογία 4 έχουμε ε, αρνητική ε, τοποθέτηση του εισηγητή. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπέρ. Ηλεκτρονική, ναι. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Η τροπολογία εγκρίνεται με 16 προς 15 ψήφους και 2 αποχές. Τροπολογία 4. Όχι, με συγχωρείτε, η 5 καλύπτεται, οπότε ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Η έκθεση όπως τροποποιήθηκε γκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ, 4 αρνητικές ψήφους και καμία αποχή. Και τώρα θα ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Σίκτριτ Μουρεσάν για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περιοχή κάποια τουρζή στη Ρουμανία με 4.000 με ε, εκατομμύρια κινητοποίηση. Ε, τροπολογία πρώτη. Δεν χρειάζεται να ψηφιστεί, καλύπτεται. 8. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 8. Κατά. αποχές μία αποχή απορρίπτεται τροπολογία 9 Ίσως ο εισηγητής θα μπορούσε να μας από την απόψη του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τροπολογία αυτή είναι του κυρίου Νεγκρέσκου και αρχικά θα έπρεπε να πούμε ότι είναι μη παρατακτή διότι προτείνει να αυξηθεί με βάση του ποσοστού πληθωρισμού το ποσό κινητοποίηση, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει βάσει του κανονισμού του Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει όμω τώρα μια συμβαστική προφορική τροπολογία, η οποία καλύπτει το μακροχρονικό διάστημα, ώστε να είναι συμβατό με του κανόνε λειτουργία του Ταμείου Προσαρμογή και έτσι πρότεινα την προφορική τροπολογία που θα λέει το εξή. Εκφράζει την ε, δυσαρέσκειά του για την μεγάλη διάρκεια των 17 μηνών και λόγω του ποσοστού πληθωρισμού στην περίοδο 2012-2014 υπήρξε μείωση τη αγοραστική δύναμη. Καλεί λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό σε παρόμοιε καταστάσει στο μέλλον. Με αυτή τη μορφή μπορούμε να το δεχτούμε. Quels sont ceux qui sont favorables à l'amendement? Υπέρ με την προφορική τροπολογία του συγκεκριτή μας κατά τρει αρνητικέ ψήφοι αποχές δεν υπάρχουν αποχές μία αποχή με την τροποφορική τροπολογία λοιπόν του συγκεκριτή μα εγκρίνεται η τροπολογία Τροπολογία 10. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Απορρίπεται. 11. Με προφορική τροπολογία του εισηγητή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με την προφορική τροπολογία προτείνουμε τη διαγραφή του τελευταίου τμήματος της τροπολογίας, Οπότε η τροπολογία λέει το εξή. Τονίζει ότι αγορά, οι συνθήκε αγορά εργασία άλλαξαν αλαφρώς τους τελευταίου 17 μήνε και πιστεύω ότι με περαιτέρω ανάλυση τη οικονομική και χρηματοπιστωτική ε, κατάσταση το 2014 θα καλύψουμε τι ανάγκε μα. Τέλο. Το υπόλοιπο τμήμα διαγράφεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα να αναθεώρηση για να μην αντίκειται η πρόβλεψή μα στου κανόνε λειτουργία του Ταμείου. Με αυτήν την εναλλαγή προτείνω να εγκριθεί η τοπολογία. Προφορο... Τροπολογία 11 λοιπόν με προφορική τροπολογία του συγγητή υπέρ. Κατά. Τρεις αρνητικές ψήφοι. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν, όπως προφορικώ τροποποιήθηκε η τροπολογία 11. 12. Ο εισηγητής είναι υπέρ, με μία διευκρίνηση, την οποία, της οποίας έχετε λάβει γνώση, υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τρεις αρνητικές ψήφοι. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Αγκρίνεται. 13. Καλύπτεται. 14. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Εννέα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 όσοι για είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Τρεις, τέσσερις, πέντε. Αποχές. Κανείς. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Θα έχουμε δυσκολία να μετρήσουμε, γι' αυτό να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Εψήφισαν άπαντες. Πέρασου. Η τροπολογία εγκρίνεται με 17 ψηφού προ 13 και μία αποχή. Τροπολογία 18. Υπέρ ο εισηγητής, υπέρ. Κατά. Αποχές. Τρεις αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποθέσεις. Απορρίπτεται. Τροπολογία πρώτη. Καλύπτεται. Το ίδιο και η δεύτερη. Τροπολογία τρία. Υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία τέταρτη. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας. Η τροπολογία εγκρίνεται με 16 προς 13 ψήφους και τρεις αποχές. Τροπολογία 5. Ο εισηγητής είναι κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρα Η τροπολογία εγκρίνεται με 16 προς 13 ψήφους και 3 αποχέ. Τροπολογία 6 καλύπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Να ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας. Το τροποποιημένο κείμενο εγκρίνεται με 29 ψήφους προς 3. Χωρίς αποχές. Και τώρα καταλήγουμε στο σχέδιο έκθεσης της Ανελή Γιάτενμάκη Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την περιοχή της Αραγώνας Τροπολογία 6 αυτή όμως καλύπτεται Υπάριθμον 7 με μια υποτροπολογία που βρίσκει σύμφωνη την εισηγήτρια υπέρ κατά αποχές ούτε κατά υπάρχουν ούτε αποχές υπαριθμών 8 υπέρ η εισηγήτρια υπέρ κατά. Τρεις ψήφοι κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν. Τροπολογία 9. Σχέτια σύμφωνη υπέρ. Κατά δεν υπάρχουν κατά. Α, υπάρχει μια ψήφος κατά. Αποχές. Όχι. Υπαριθμόν 10. Η συγγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 11. Εδώ υπάρχουν δύο διευκρινήσεις με μορφή τροπολογιών. Πρώτη, ψηφίζουμε σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος, εκεί είναι σύμφωνη η συγγήτρια, υπέρ, ψήφι υπέρ δηλαδή, κατά, αποχές, δεν υπάρχουν αποχές. Για το δεύτερο μέρος τώρα, εκεί που λέει points out κλπ. Η, η εδώ είναι αντίθετη, ψήφι υπέρ. Ψηφίστε παρακαλώ με, ηλεκτρονικές, με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε άπαντες. Τέλος. Άρα το δεύτερο μέρος εγκρίνεται με ψήφους 17 υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 12. Πάλι εδώ είναι δύο μέρη, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, η εισηγήτρια είναι υπέρ, ψήφι υπέρ. Ομοφόνος. μία ψήφος κατά και μία αποχή. Καλά. Για το δεύτερο μέρος, εδώ η εισηγήτρια είναι αντίθετη, υπέρ, ψήφι υπέρ. ψήφι κατά. Έξι ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν και το δεύτερο μέρος. Τροπολογία 13. Η συγκήτρια υπέρ. Η ψήφι υπέρ. Κατά. Τη ψήφι κατά. Αποχές δεν υπάρχουν. Τροπολογία 14. Η δεν είναι υπέρ. Ψήφι υπέρ. Κατά. Ψήφι 3 κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. 16. Η υπέρ. Υπέρ. Ψήφι υπέρ. ψήφι κατά, ούτε αποχές. 16, η χειρίτρια είναι υπέρ. Κατά, παρακαλώ. Δεν υπάρχουν αποχές. Τροπολογία 17. Εδώ υπάρχει μια υποτροπολογία της ίδιας της ηγήτριας στην οποία δίνω το λόγο. Α, δεν είναι, παν, δεν είναι παρούσα, μάλιστα. Καλά. Γνωρίζετε πάντως την τροπολογία της τώρα. Και με την επιφύλαξη τώρα αυτής της υποτροπολογίας έχει εκφράσει θετική γνώμη. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Τέσσερις κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Τροπολογία 1 έχει καλυφθεί, η 2 ομοίως, η 3 όπου είναι υπέρ, η εισηγήτρια ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν και τροπολογία 4. Πάλι εδώ είναι υπέρ η εισηγήτρια ψήφι υπέρ. Μου φαίνεται ότι θα είναι ομόφωνα υπέρ. Η ψήφος δεν βλέπω ούτε αποχές. Άλλωστε η παριθμόν 5 καλύπτεται. Άρα θα ψηφίσουμε τώρα το κείμενο στο σύνολό του ως ετροποποιήθη και αρχίζει η ψηφοφορία ηλεκτρονική. Ψηφίσατε άπαντες πέρας της ψήφου η δε έκθεση όσο τροποποιήθη υπερψηφίζεται με ψήφους 29 υπέρ και 3 κατά και καμία αποχή. Τώρα εδώ ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεπρέ για 7 μεταφορές πιστώσεων που, όπου απαιτείται θετική γνώμη της Επιτροπής μας. Πρόκειται για το τμήμα 3, κυρίως τώρα το 30, η μεταφορά πιστώσεων 30 που αναφέρεται στο Νότιο Σουδάν έχει σημασία. Ο κ. Ντεπρέ, κύριε Πρόεδρε, απλά είναι εδώ τα πράγματα υπαριθμών 12, 13, 14, 15, 16 και 17 είναι απαραίτητο να ψηφιστούν, διότι αν δεν ψηφιστούν, κάθε απόφαση που θα εγκρίνουμε δεν θα είναι δυνατόν να, καταστούν, να καταστεί λειτουργική. Άρα πρέπει να εγκριθούν οι αναγκαίες αυτές τις μεταφορές πιστώσεων στον προϋπολογισμό, έτσι ώστε οι αποφάσεις που θα λάβουμε να μπορούν να εκτελεστούν. Προτείνω λοιπόν, εάν δεν υπάρχει ένσταση, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί, διότι ακολουθούν όλες την ίδια λογική. Και μετά θα διακόπτει ο Πρόεδρος. Άρα λοιπόν για τις έξι τροπολογίες, δεν είναι τροπολογίες, πρόκειται για μεταφορές πιστώσεων. Μάλιστα για τις έξι μεταφορές πιστώσεων και τροπολογίες. Στην ουσία αυτές αποτελούν την τη συνέπεια της ε, ψήφου που διεξάγαγαμε. Και επομένως θέτω σε ψηφοφορία όλες μαζί τις μεταφορές αυτές πιστώσεων. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η αντίθετη ψήφι. Η αντίθετη ψήφι. Τρεις ψήφοι κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. Α, υπάρχουν δύο αποχές. Κύριε Ντεπρέ, λαμβάνετε το λόγο για την υπαριθμό 30. Όπως είπατε πριν, Πρόκειται για κατεπίγουσα αίτηση, πρόκειται για 20 εκατομμύρια ευρώ και για υποχρεώσεις και για πληρωμές από το αποθεματικό ανθρωπιστικής βοήθειας κατεπίγοντος χαρακτήρα για επισητιστική βοήθεια και αντιμετώπιση θεομηνιών. Για να προσφερθεί βοήθεια στα θύματα των ε, συγκρούσεων στο νότιο Σουδάν, με, στα οποία περιλαμβάνεται μάλλον μεγάλος αριθμός παιδιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει, ήθελε μάλλον ήδη από τον Αύγουστο να εισαγάγει τη σχετική αίτηση, λόγω όμως της συμφωνίας που έγινε, δεν μας ζήτησαν να εργαστούμε Αύγουστο μήνα, πάντως όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι κατεπίγονο χαρακτήρας και παρακαλώ να υπερψηφιστεί. Ο Πρόεδρος, επιθυμεί κανείς να λάβει το λόγο. προτείνει ο κύριος Ντεπρέ να υπερψηφίσουμε τονίζοντας και τον κατεπήγοντα χαρακτήρα. Θέτω σε ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ. Νομίζω ότι σηκώθηκαν πράγματι όλα τα χέρια. Δεν υπάρχουν ψήφοι κατά, ούτε αποχές. Καλά λοιπόν, θα τελειώσουμε. Μάλλον τελειώνουμε εδώ την ψηφοφορία. Ίσως βιάστηκα να το πω προηγουμένως. Όταν δηλαδή ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία για τις ε, Τροπολογίε για την έκθεση για το Ταμείο παγκοσμιοποίηση. Τώρα, προπολογισμό 2015 έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η φάση της καταθέσεως τροπολογιών. Ελπίζω ότι ήταν γόνιμη. Οι προθεσμίε για τις πολιτικές ομάδες ε, λήγουν σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γενική Εισηγήτρια Γάρδια Ζαμπάλ για να εξηγήσει θα δώσω μετά το λόγο στους ε, βουλευτές που επιθυμούν να τον λάβουν. Η κυρία Γενική Συγκήτρια. Sí, muchas Ευχαριστώ. Όπως είπατε και εσείς σωστά, έχουν κατατεθεί κάποιες πρώτες τροπολογίες και σήμερα εκπνέει η προθεσμία οι τροπολογίε φυσικά σχετίζονται με τις προτεραιότητε των ε, βουλευτών. 890 ε, ήταν οι αρχικέ τροπολογίε, 515 από τις ε, συναρμόδιες επιτροπές και 365 από μεμονωμένου βουλευτέ. Είναι αρκετά υψηλό ο αριθμός των τροπολογιών, όμως εάν συγκρίνουμε με άλλες διαδικασίε έγκριση προπολογισμού δεν είναι τόσο υψηλός ο αριθμός των τροπολογιών. Υπάρχει ορισμένες φορές για τους προϋπολογισμούς που είναι ανάμεσα σε δύο ε, περιόδους, ε, οικονομικές περιόδους, ε, προκύπτουν και οργανωτικής φύσης προβλήματα, προβλήματα υποβολής, παρουσίας των τροπολογιών και είναι φυσιολογικό ανάλογα και με τον αριθμό προτεραιοτήτων να αυξάνεται και ο αριθμό των τροπολογιών. Λοιπόν, ας δούμε τις δαπάνε σε ανακατηγορία. Ένα α, ανάπτυξη, απασχόληση, καινοτομία. 192 ε, ήταν συνολικά οι τροπολογίες ε, σε αυτήν την κατηγορία για όλες τις κατηγορίες εξάλλου. Η ε, κατεύθυνση που ακολουθούν οι είναι η επαναφορά της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ούτως ώστε ως προς πιστώσεις που χρειάζονται και τις πιστώσεις πληρωμών τελικά ε, να καταργηθούν, να αναιρεθούν οι περικοπές που μας προτείνει το Συμβούλιο. Ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, για το Εράσμους, για τις κοινωνικές ε, επιχειρήσεις. Υπερβαίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης προτείνουμε αύξηση των κονδυλίων για τις υποπτικές αρχές, όπως και τα προηγούμενα έτη, για πιλωτικές δράσεις και προπαρασκευαστικές δράσεις. Επίσης υπάρχουν κάποιες τροπολογίες. Αν δούμε τώρα πόσες υπερβαίνουν ε, της αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τελικά ε, την εξεπερνούμε με 62 ή 63 εκατομμύρια για την κατηγορία 1β για τα διαρθρωτικά ταμεία και τις περιφερειακές πολιτικές 33 συνετροπολογίες ο στόχος είναι η επαναφορά της αρχικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και με πολλές τροπολογίες ε, αποσκοπούν στην αύξηση των κονδυλίων γιατί εκεί εντοπίζονται και οι περισσότερες δυσκολίες. Ο στόχος είναι να περατωθούν δε τα προγράμματα που έτρεχαν ε, στο προηγούμενο πολιετές σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίση, υπάρχει η πρόταση για αύξηση του Ταμείου για τους Πλέον Απόρους. Είναι ένα πρόγραμμα που ε, έχει ιδιαίτερε δυσκολίε για τι ανάληψη υποχρεώσεων. Προτείνουμε αύξηση κατά 22 εκατομμύρια και επίση υπάρχει μια άλλη τροπολογία για την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών. 9 εκατομμύρια ε, για, τις, ε, για την ανάληψη υποχρεώσεων και 7 για τι πληρωμέ. και όπω έλεγα, οι περισσότερε τροπολογίε είναι για την επαναφορά τη αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν όμω και τρει ε, τροπολογίε που ε, ζητούν 200, 250 εκατομμυρία για μία γραμμή για τη ζάχαρη και την αναδιάρθρωση ε, του κλάδου. Επίση, 3 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια ζητούνται σε μία άλλη τροπολογία. Είναι μία επιτροπή περιβάλλοντο, Είναι εξαιρετικά φιλόδοξη οι συνάδελφοι που κατέθεσαν τροπολογία για τα 3 δις 200 εκατομμύρια ζητούν αλλαγή των πυλών. δηλαδή να περάσουμε από τις άμεσες ενισχύσεις στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Ε, στην κατηγορία 3 είχαμε στο σύνολο 66 τροπολογίες, η πλειοψήφια και πάλι είναι για ε, επαναφορά της αρχικής πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροφής. Το πρόγραμμα Creative Europe και η δράση για τα πολυμέσα. Έχουμε διάφορους οργανισμούς για την καταπολέμηση ε, της ε, τοξικομανίας Frontex ε, και διάφοροι άλλοι οργανισμοί. Ο στόχος είναι αύξηση κατά 20 δις του προϋπολογισμού ε, διατηρώντας και ένα αποθεματικό ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν κατεπηγόντως χρειαστούν κονδύλια, θα είναι ήδη γεγραμμένα στην αντίστοιχη γραμμή και θα κινητοποιούνται ως ε, εκ τούτου εύκολα, μετά φυσικά από την ε, συγκατάθεση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε δηλαδή σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που θα είναι πολύ πιο χρονοβόρα η διαδικασία. Αν προκύψει ε, η ανάγκη στην κατηγορία 4, όπως και στην 1α, έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες, 147 το αριθμό και 392 ε, εκατομμύρια. Αυτή είναι η αύξηση που ζητούμε σε σχέση με την πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ ξεπερνούμε τα διαθέσιμα περιθώρια. Αν είναι να δεχτούμε ε, το σύνολο θα χρειαστεί να προσφύγουμε στο μέσο ευελιξίας ε, διότι το έλλειμμα ανέρχεται πλέον στα 56 εκατομμύρια αν εγκριθούν όλα αυτά. Ε, οι προτεραιότητες τώρα των αρμοδίων επιτροπών ε, έχουν ε, ιστορική σημασία στο Κοινοβούλιο. Πρόκειται για τη βοήθεια προς τους Παλαιστινίους, βοήθεια προς τις νότιες και ανατολικές χώρες. Στην κατηγορία 5 έχουμε 22 τροπολογίες για την ανέρεση των περικοπών που εισηγείται το Συμβούλιο για τα διάφορα προγράμματα. Αναφέρθηκα ακροφυγώς και στους οργανισμούς. Ε, συνοψίζοντας το τι συνέβη με αυτούς τους οργανισμούς, για 15 από αυτούς τους οργανισμούς περιέκοψε τα κονδύλια το Συμβούλιο, για τους 8 από, από τους 15 αποκαταστάθηκε ο προϋπολογισμός και για, τις, ε, για τους 6 με τις τροπολογίες που καταθέτουμε υπερβαίνουμε την αρχή πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφήστε που έχουμε δύο είδη τροπολογιών. Οι μεν προτείνουν αύξηση των κονδυλίων για τους οργανισμούς, οι δε προτείνουν τροποποίηση του οργανογράμματος των οργανισμών, διότι ξέρετε πως ε, στην Επιτροπή υπήρξαν δύο φάσεις προσαρμογής για τους οργανισμούς ε, Πρώτον, ε, μείωση κατά 5% ε, του προσωπικού και 1% των κονδυλίων για μία πενταετία και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, ε, πρόταση δημιουργίας μιας, ενός αποθέματος ανθρωπίνων πόρων για έκτακτες ανάγκες. Το Κοινοβούλιο δεν συμφωνεί ε, να ε, περικοπούν τα 5% σε σχέση με τα 5%, το 5% που ήδη είχε εγκριθεί. Αν κάνουμε μια αντιπαράθεση του οργανογράμματος με το προηγούμενο 5%, καταλαβαίνετε ότι μπλέκονται τα πράγματα γιατί έχουμε το αρχικό 5% και το ε, πρόσθετο 5% και άρα δύσκολο μπορεί να σχηματίσει κανείς μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτά προτείνουν οι συναρμόδιες επιτροπές και τώρα θέλω να ξέρω τι προτείνουν οι πολιτικές ομάδες. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία, όπως είπαμε. Θέλω όμως να γνωρίζω ποιε είναι οι πολιτικές προτεραιότητες των πολιτικών ομάδων για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Θα πρέπει να Γνωρίζουμε επίσης πως οι επιδιωκόμενοι στόχοι για τις για τη στρατηγική, για τις επιστώσεις πληρωμών και για τις προτεραιότητες ε, που θα κληθούμε να υλοποιήσουμε σχετίζονται και με την ε, ε, ε, πληρωμή των ανεξόφλητων λογαριασμών των καθυστερούμενων ε, πληρωμών, ε, γιατί είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις που σημειώνονται. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την Γενική Συγγήτρια τώρα. Ε, ας ακούσουμε συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Φερνάντες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή, νομίζω τουλάχιστον, ε, δεν αρχίζουμε συζήτηση για τις ε, τροπολογίες ε, αυτές καθ' αυτές. Φυσικά για τις γραμμές και τις προτεραιότητες που έχουμε συμφωνούμε, συμφωνούμε για την κατηγορία 1α, για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ε, θεωρούμε ότι υπάρχει ένα προσεπίληση πρόβλημα και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το ε, επιλύσουμε ή να το ελαχιστοποιήσουμε τουλάχιστον για το 2015. Είναι φυσικά το πρόβλημα των πληρωμών. Δεν μπορούμε να λησμονήσουμε ότι το πολιετές δημοσιονομικό που εγκρίναμε από το 2014 έως το 2020 είναι κατώτερο του προηγουμένου 2007-2013 και το Κοινοβούλιο ως εκ τούτου ζήτησε μέσω ευελιξίας. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε λοιπόν την απόφαση για την αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού ε, και μέχρι το 2016 αναμένεται πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Λοιπόν, Πρέπει να είναι αξιόπιστος ο προϋπολογισμός μας. Πρέπει να συμμορφωθούμε με την ε, νομοθεσία. Δεν μπορούμε να χρωστάμε. Ε, γι' αυτό και είναι τόσο επίγον αυτό το πρόβλημα των ε, πληρωμών για τον προϋπολογισμό 2015. Πέραν αυτού είναι απαράδεκτο που το Ταμείο για την υποστήριξη προς τους πλέον απόρους να προ προς τα κονδύλια του. Τα κοινωνικά θέματα, ε, οι τροποποιήσεις για το γάλα και για τα φρούτα ε, στα σχολεία ε, είναι θέματα και ε, αντικείμενα των τροπολογιών που πιστεύω όλοι θα υποστηρίξουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πέρα από τα προβλήματα, την, ε, εκτός από την εσωτερική αλληλεγγύη και την εξωτερική αλληλεγγύη με την αναπτυξιακή βοήθεια, κατηγορία 4, προβλήματα γειτονία, θέματα που σχετίζονται με την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι προφανές ότι και αυτές οι τροπολογίες θα τύχουν συνολικής υποστήριξης τουλάχιστον από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ήθελα μόνο να υποστηρίξω τον τα αυτά που είπε για την ανθρωπιστική βοήθεια. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους δωρητές λόγω των περικοπών περιμένουν ακόμη οι αρμόδιοι τα 10 εκατομμύρια που έπρεπε να έχουν ήδη πληρωθεί τον προηγούμενο μήνα και είναι προφανές ότι ε, αντιμετωπίζουν σοβαρή κρίση γιατί έχει και παράπλευρες επιπτώσεις όλες οι υπηρεσίες ε, που μπορούν, ε, προσπαθούν να προσφέρουν επιτόπου. Θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε κάποια θέση ούτως ώστε να εκταμιευθούν τα υπεσχημένα οι πληρωμές και να ιεραρχήσουμε τις ε, προτεραιότητες. Ε, δηλαδή, ε, ποια, ποια είναι κατεπήγοντα, ποια πρέπει κατεπήγοντας να πληρωθούν. Σε κάθε περίπτωση, όλα, εντάξει, όταν έχουμε ανθρωπιστική κρίση, όλα επίγοντα είναι, αλλά σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον για την καθαρά ανθρωπιστική βοήθεια, πρέπει να ιεραρχήσουμε αυστηρά τις προτεραιότητες. Ευχαριστούμε, Σανή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς συμφωνούμε απολύτως να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, το σοβαρότερο το πρόβλημα με τις πληρωμές και Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει προτεραιότητες. Έχουμε προϋπολογισμό, έχουμε προβλέψει κάποια κονδύλια και εντός αυτών των κονδυλίων θα πρέπει να δούμε από πού μπορούμε να πάρουμε κάποιους πόρους για να τους μεταφέρουμε προς τις προτεραιότητες που έχουν θέσει το Κοινοβούλιο και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη φωνή του Προέδρου της, του κ. Γιούνκερ προτεραιότητες που καθορίστηκαν για ολοκληρή τη θητεία της. Η ανεργία των νέων, η ανάπτυξη και το κεφάλαιο 3 κυρίως για τη μετανάστευση. Προτείναμε λοιπόν σχετικά κάποιες τροπολογίες για να αλλάξει και το κονδυλί που προβλέπεται για τη Frontex και το πρόβλημα με τις μετανάστευσεις να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να αναλάβει ευθύνη ολόκληρη η Ευρώπη για αυτό το ζήτημα. Όσο για το 5 Στο κεφάλαιο 5 καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προσπάθειες για να εντοπίσει ποιες δαπάνες είναι δαπάνες προτεραιότητας. Κατά την άποψή μας, εδώ υπάρχει περιθώριο ε, περαιτέρω παρέμβασης για να δούμε αν μπορούμε να μεταφέρουμε κάποιους πόρους προς ε, άλλα σημεία του προπολογισμού σε προτεραιότητες που θεωρούμε πιο επίγουσες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο, στην ομάδα μας δεν έχει ολοκληρωθεί σχετική συζήτηση. Αλλά θα σας αναφέρω σε ποια σημεία συμφωνούμε ήδη. Θεωρούμε κατά πρώτο για τον προϋπολογισμό και για την εκτέλεση του προπολογισμού 2014 και για τον προπολογισμό το 2015 θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις πληρωμές. Η τρέχουσα κατάσταση είναι αρκετά ανησυχητική. Δεν είναι εύκολο να ε, την αντιμετωπίσει κανείς αν συνεχίσει το Συμβουλίο να βρίσκεται στην ίδια θέση και να ε, μεταβάλει τη στάση του. Έχουμε ελάχιστε πληρωμές αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε τα αρχικά ποσά που προέβλεπε η Επιτροπή. να γίνουν κάποιες προσαρμογές μεταξύ διαφορετικών τίτλων και προβλεπόμενων πιστώσεων ε, στις γραμμές του προπολογισμού. Για τις υποχρεώσεις τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση, αλλά έστω για το επίπεδο των ε, υποχρεώσεων είναι ανεύθυνο να ζητούμε να επιληθεί το ζήτημα των πληρωμών εάν προηγουμένως δεν έχει επιληθεί το ζήτημα των υποχρεώσεων. Εάν δεν ε, αλλάξει η σκοπιά μας ως προς τις υποχρεώσεις θα εξακολουθήσει και το πρόβλημα με τις πληρωμές. Θα επιδεινωθεί δηλαδή στο μέλλον. Πρέπει να δούμε το επίπεδο των υποχρεώσεων και εκεί να σκεφτούμε πού θέλουμε να φτάσουμε για το 2015. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητε και το περιθώριο ελιγμού που έχουμε στον προπολογισμό για το 2015 και ανάλογα με το ανώτατο όριο, το οποίο θα φτάσουμε στις υποχρεώσεις, θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες για την κατάσταση της Ανατολικής Ευρώπης, ιδίως για την Ουκρανία όπου έχουμε ιδιαίτερες ευθύνες ενώπιον της χώρας αυτής και δεν μπορούμε να δεχτούμε το κράτος αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι θύμα ενός υπόγειου πολέμου και οικονομικής κρίσης να μην μπορέσει να ξεφύγει από αυτή. Επίσης, θεωρούμε ότι το ύψος των πιστώσεων για την ανθρωπιστική βοήθεια και τις κατεπήγουσες ε, συνθήκες, ιδίως στη Μέση Ανατολή την Αφρική, θεωρούμε ότι τα ποσά αυτά θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να αυξηθούν. Κατά τρίτον, παραδοσιακά ξέρετε ότι προσοχή δίνουμε στο σύνολο των προγραμμάτων που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξυγχρονιστούν και να συμμετέχουν καλύτερα στην αγορά και τέταρτον δίνουμε μεγάλη σημασία στην ενίσχυση αυτού που αποκαλούμε ψηφιοποίηση. Δηλαδή ψηφιακή οικονομία. Λίγο πολύ από τις διάφορες δημοσιονομικές γραμμές αυτό είναι το σύνολο των προτεραιοτήτων μας για τον προπολογισμό το 2015. Πρόεδρος, ευχαριστώ, ο κύριος Κόλμπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα ευχαριστώ την ίδια την εισηγήτρια. Άκουσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι δεν τρομάζει καν απέναντι στις χίλιες τροπολογίες. Μπράβο, τη συγχαίρω. Εμείς της ομάδα CCR συζητήσαμε την εβδομάδα αυτή τον προϋπολογισμό. Οφείλω δεν να σας πω ότι θα τον απορρίψουμε τον προϋπολογισμό, διότι σε αυτόν δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται το θεμελιώδες πρόβλημα αυτή τη όλο και μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ πιστώσεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών. Κάτι για το οποίο έχουμε ήδη μιλήσει. Νομίζω δεν χρειάζεται να επεκταθώ περισσότερο σήμερα. Αυτό το πρόβλημα το βλέπουμε και μάλιστα απόλυτα ξεκάθαρα το βρίσκουμε ότι είναι και πρόβλημα νομικής φύσης διότι από αυτές τις πιστώσεις υποχρεώσεων που δεν καλύπτονται μπορεί κάποια στιγμή να καταλήξουμε σε χρέη. Και χρέη δεν επιτρέπεται να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο γνωρίζετε. Έχουμε λοιπόν ορισμένες τροπολογίες που έχουμε καταθέσει ως πολιτική ομάδα, διότι θεωρούμε ότι σε ορισμένα σημεία μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις χρημάτων, μπορούν δηλαδή ορισμένα χρήματα να δαπανηθούν καλύτερα, κυρίως όταν πρόκειται για επενδύσεις για ανάπτυξη και απασχόληση Ασφαλώς αυτά είναι αδιαμφισβήτητα, τα είπαν και άλλοι που μίλησαν πριν. Έτσι λοιπόν, θέλουμε μια ισχυρότερη στόχευση προς τους τομείς αυτούς. Για αυτό το λόγο έχουμε κάνει και σχετικές τροπολογίες που ανέρχονται σε περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ και που θεωρούμε ότι μπορούν να εξοικονομηθούν τα χρήματα αυτά για να μπουν σε αποθεματικά. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ντεζανού. Η συζήτηση αυτή είναι ενδιαφέρουσα. Αλλά όσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ορίζει αυτό τα έσοδα, στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να ανοίγουμε τρύπες για να καλύψουμε άλλες. Πρέπει άρα να καθορίσουμε προτεραιότητες. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν τρεις ξεκάθαρες προτεραιότητες. Πρώτη, τα ανθρωπιστικά και τα θέματα αλληλεγγύης με κάθε άποψη, και εσωτερικά και εξωτερικά. Δεύτερο, Βεβαίως η ανάπτυξη και η απασχόληση. Και αυτά μάλιστα συνδέονται. Και τέλος ως πρόεδρος περιφέρειας δεν μπορώ να λησμονήσω τα διαρθρωτικά ταμεία. Πολλές κοινότητες, τοπικές διοικήσεις αναμένουν τα χρήματα αυτά για να βρεθούν κάποιες λύσεις. Νομίζω ότι το ζήτημα των πληρωμών είναι ασφαλώς ζήτημα προτεραιότητας και πρέπει εκεί να δράσουμε όλοι μαζί για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Ξαναλέω ωστόσο ότι πρέπει να εξευρεθούν νέοι πόροι αν θέλουμε να μπορέσει πραγματικά η Ευρώπη να έρθει στο ύψος των υποχρεώσεών της για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τεσόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνει το λόγο. Ευχαριστώ και σας συγχαίρω που είπατε τόσο σωστά το όνομά μου. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την θαυμάσια εργασία που έχει επιτελέσει για το σχέδιο του προϋπολογισμού. Ο ίδιος εγώ προσωπικά ως εισηγητής για λογαριασμό της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι το έργο της σύνταξης του σχεδίου προπολογισμού και γι' αυτό πραγματικά της βγάζω το καπέλο. Από τη δική μου άποψη είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην χρεωθεί, να μην αναλάβει χρέη. Πρέπει να φανούμε υπεύθυνοι και πρέπει να είμαστε σόφρονες και προβλέψιμοι. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες κυρίως δε των ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών, έχουν μεγάλη αγωνία για το μέλλον και φοβούνται και για την ίδια την ασφάλειά τους. Εγώ θα επανέλθω σε αυτά που είπαν προηγούμενοι ομιλητές. Η ασφάλεια, η μετανάστευση, αυτά είναι πράγματα όπου δεν πρέπει να κάνουμε εξοικονομήσεις. Ωστόσο πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού μελετώ προσεκτικά έναν αριθμό προγραμμάτων και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν τρόποι να γίνουν εξοικονομήσεις, όχι για τα ανθρωπιστικά, αλλά σε ορισμένα άλλα προγράμματα όπου έχουν σπαταληθεί χρήματα, διότι πολλά χρήματα έχουν σπαταληθεί. Διοργανώνονται συνέδρια ως αυτός σκοπός. Ξεκινούν έργα τα οποία δεν έχουν επιλεχθεί επειδή είναι τα καλύτερα αλλά μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν ορισμένες χώρες μέλη. Εγώ λοιπόν θα αντιταχθώ σε οποιαδήποτε κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η συζήτησή μας για τον προϋπολογισμό στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι διαφορετική από αυτήν που γίνεται οι δημοσιονομικές συζητήσεις δηλαδή στις χώρες μέλη. Διότι μιλούμε για πρόγραμμα. Τι θα πρέπει να κάνουμε. Έχουμε χρήματα για να τα κάνουμε αυτά που θέλουμε. Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε προτεραιότητες ανάλογα με τα χρήματα που διαθέτουμε ή πόσα χρήματα χρειαζόμαστε για να ικανοποιήσουμε τις προτεραιότητες. Αυτά είναι για το προγραμματισμό των επόμενων ετών. Εμείς όμως βρισκόμαστε τώρα σε ιδιαίτερη κατάσταση, διότι καλούμεθα να συζητήσουμε το πρόγραμμα των εργασιών, χωρίς να γνωρίζουμε ωστόσο πόσο μεγάλο θα είναι το χρέος. Αυτό θεωρητικά βέβαια, διότι δεν θα έχουμε. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα ελλείμματα μέχρι τέλους του 2014. Μπορούμε βέβαια να προβλέψουμε πάνω κάτω σήμερα, τώρα τον Σεπτέμβρη, μόνο στον τίτλο 1β το κενό σήμερα ανέρχεται στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. 10 δις περίπου. Επομένως, οι αξιώσεις που έχουν φτάσει, οι απαιτήσει που έχουν φτάσει τώρα και περιμένουν πληρωμές ανέρχονται στα 10 δις και μας μένουν 3, 3 μήνες ακόμα μέχρι τέλους του έτους. Με πολύ ενδιαφέρον λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί το έλλειμμα αυτό μέχρι τέλους του έτους μπορούμε να το υπολογίσουμε λίγο πολύ. Άρα ανατρέπεται η κατάσταση αυτή. Δηλαδή δεν μπορούμε τώρα να προγραμματίσουμε διότι δεν ξέρουμε πόσα λεφτά πρέπει να δώσουμε για τις παλιές, για να ξεπληρώσουμε τις παλιές υποχρώσεις. Και εμείς ξεχνούμε ότι το 2015 είναι ο τελευταίος, ε, η τελευταία χρονιά του νη συν 2. Και επομένως εκεί λήγουν όλα τα προγράμματα της περίοδου 2007-2013. Αυτό όμως σημαίνει ότι ο προπολογισμό μας για το 2015 σύμφωνα με τις οροφές που έχουμε, γιατί οι οροφές είναι αυτέ που το καθορίζουν, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα και πρέπει να το έχουμε υπόψη μα αυτό. Δηλαδή όσο συζητούμε το 2015 δεν έχουμε λύσει ακόμα το πρόβλημα. Θα εξακολουθούμε να έχουμε ένα μεγάλο κενό στον προπολογισμό. Για να είμαστε τώρα λοιπόν απόλυτα ειλικρινεί, αυτό που κάνουμε εμεί στην πραγματικότητα είναι ότι προσπαθούμε να επιδιορθώσουμε το σύστημα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει να αλλάξει το σύστημα. Και προτείνονται διαφορετικέ λύσει ανάλογα με διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσει. Τι γίνεται όμω με τι υποχρεώσει που πάνε πίσω στους καθαρούς συνεισφορείς. δεν πληρώσουμε τις αξιώσεις, δεν πληρώνουμε μάλλον τις, ε, δεν ξεπληρώνουμε δηλαδή τις ανηλμένες υποχρώσεις μας, παρόλα αυτά δίνουμε λεφτά πίσω στις χώρες μέλη. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Προσπαθούμε να κάνουμε να επιδιορθώσουμε το σύστημα όπως είπα, χωρίς να γνωρίζουμε ωστόσο ποια είναι η πραγματική κατάσταση του προπολογισμού τελικά. Εννοώ το, το, έλλειμμα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι, να συγχαρώ την ε, κύριε Συγγετρία για τον προπολογισμό. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι η όλη διαδικασία. Το πρόβλημα όμως που βλέπουμε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να δυστυχώς είναι το ίδιο ε, κάθε δημοσιονομικό έτος. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία μεταβολή στην χάραξη πολιτικής Ιδίω ω προς τον προπολογισμό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έπρεπε να υπάρξει κάποια αναθεώρηση του προπολογισμού, ώστε οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προ τα κάθε μέλη να καλύπτονται, αν μη τι άλλο. Αυτό, από μόνο του, δημιουργεί μεγάλα ελλείμματα στα κράτη-μέλη. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων και συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να κάνει διάλογο και να συζητήσει και τον προπολογισμό όπως εγκρίθηκε από το όπως θα εγκριθεί μάλλον από το Ευρωκοινοβούλιο. διότι πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με το τι συμβαίνει στην πράξη διαρκώς παραβια... παραβαίνονται οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν καλύπτονται τα χρέη που δημιουργούνται. Υπάρχει και ο περιορισμός του 3% για το κρατικό έλλειμμα και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν καλύπτει τις υποχρεώσεις της προς τα κάτι μέλη, δεν καταβάλει τις πληρωμές της. Κύριε Πρόεδρε, προτείνατε ε, προτάθηκε μάλλον και ακούστηκε η ιδέα, ίσως να έρθουμε σε επαφή με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές επί των προπολογισμών από τα κράτη-μέλη. Ίσως έτσι να βρούμε κάποια λύση και να φανούμε πιο ευέλικτοι στις ιδέες που θα σκεφτούμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Θα προσφέρουμε έτσι υπηρεσία και στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρκεί απλώς η γνώμη των υψηλά ιστάμενων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από ό,τι φαίνεται. Ευχαριστούμε. Κυρία Εισηγήτρια, θα πρέπει να αισθάνεστε μεγάλη ανακούφιση μετά τις παρατηρήσεις που μόλις έγιναν. Θα μπορέσετε ίσως να ιεραρχήσετε καλύτερα έτσι τις διάφορες τροπολογίες και να δώσετε κάποια μεγαλύτερη έμφαση σε ορισμένες σε σχέση με άλλες. Ευχαριστώ πάντως όλους τους συναδέλφους για αυτές τους, τις τοποθετήσεις. Νομίζω ότι έτσι μπορείτε να καθορίσετε καλύτερα κριτήρια επιλογής. Ε, κυρία Συγκέντρια, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Και να πω ότι νομίζω ότι ως προς τις πιστώσεις υποχρεώσεων και για να να καλυφθούν και τα σχόλια των ε, συναδέλφων, νομίζω ότι θα βρούμε κάποια πολιτική συμφωνία ε, με τις προτεραιότητες που έχουμε καθορίσει όλοι ως προς τις υποχρεώσεις. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει με το Συμβούλιο είναι αυτό των πληρωμών πώς θα γεφυρώσουμε την, το χάσμα, την μεγάλη απόσταση μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών. Τα εργαλεία που διαθέτουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα είναι κάπως περιορισμένα. Υπάρχει ένα περιθώριο 4 δις ευρώ, τα οποία μπορούμε να κινητοποιήσουμε, αλλά αυτό δεν καλύπτει το κενό των 23 δις από το 2013, ούτε όλα τα πλήρωτα από που θα έχουμε το 2015. Νομίζω λοιπόν το πρώτο συμπέρασμα στο που μπορούμε να καταλήξουμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτή είναι η προτεραιότητα για την Επιτροπή μας και θα το συζητήσουμε εντός ολίγου όταν ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για τα σημεία αυτά. Πώς θα αναθεωρηθεί τώρα το δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει αυτό. Είτε θα μειώσουμε τις υποχρεώσεις ή τουλάχιστον θα καλύπτουμε τις ε, πληρωμές. Ε, αυτά που δεσμευτήκαμε να πληρώσουμε δηλαδή θα τα πληρώνουμε. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, γιατί να αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις. Θα πρέπει δηλαδή να λαμβάνουμε υπόψη και το 1% του ΑΕΠ, το όριο αυτό, αλλά το θέμα είναι πού θα βρούμε αυτά τα 23 δις που μας λείπουν. Τι θα γίνει με τα διαρθωτικά ταμεία, την ε, πολιτική συνοχή, τι θα γίνει με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Εδώ μιλάμε για ε, δις όχι απλώς εκατομμύρια. Και σε πρώτη φάση μας λείπουν 500 εκατομμύρια. Είναι λοιπόν περισσότερο θέμα υποχρεώσεων και στάσεις του Συμβουλίου. Ακόμη και αν ε, αναλάβουμε κάποιες δεσμεύσεις, δεν θα καταφέρουμε νομίζω να λύσουμε το πρόβλημα σε μόνιμη βάση. Βλέπουμε διαρκώς να επαναλαμβάνεται αυτή η δυσκολία με τις πληρωμές. Και υπάρχει και μια διαρκή στάση να μειώνονται οι συνεισφορές προς τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Από πού λοιπόν θα περικοπούν αυτά τα 23 δις ευρώ. Δεν θα το πω αυτό εγώ ως εισηγήτρια, ούτε θα αποφασίσει η ομάδα των σοσιαλιστών αν θα αλλάξουμε την πολιτική ανάπτυξη, ε, της ανάπτυξης της υπαίθρου, την κοινή γεωργική πολιτική, ε, τις περιφερειακές πολιτικές και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε, γιατί πολλές φορές κάνουμε απλώς γενικές συζητήσεις, αλλά το περνάμε στις λεπτομέρειες, βλέπουμε ότι αυτά που ε, συζητήσαμε δεν χρησιμεύουν για να λύσουμε επιμέρους προβλήματα. Ο πρόεδρος λέει, το πρόβλημα είναι συνήθως οι λεπτομέρειες. Θα τις ξαναδούμε αυτές τις τροπολογίες και θα προσπαθήσουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις υπεύθυνε επιλέγοντας την επιλογή προπολογισμών, την Επιτροπή Προπολογισμών για Προεδρία, δείξαμε αυταπάρνηση. Αλλά θα πρέπει να φανούμε και ρεαλιστές. Στην πολιτική ο ρεαλισμός έχει πολλές φορές να κάνει με την Α, έχει να κάνει με το πώς θα αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα θέματα. Θα πρέπει λοιπόν να φανούμε κι εμείς συνεπείς ώστε να μην ε, βρεθούμε ε, χωρίς να ακουστεί η άποψή μας. Τη στιγμή που αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις και τη στιγμή που γίνονται εκταμιεύσεις, σίγουρα υπάρχει μεταξύ τους μία απόσταση. Ε, μπορεί να μεσολαβεί και ένα έτος, δύο χρόνια δεν είναι πολιτικά υπεύθυνη στάση να λέμε θα αναλάβουμε λίγες περισσότερες δεσμεύσεις λόγω χάρη υποχρεώσεις. Από, 2000, από το 2014 έως το 2020 φαίνεται να υπάρχει μία απόσταση 52 δις. Ε, δεν... Ε, Υπάρχει λοιπόν ε, συνέπεια εδώ. Έχουμε ένα πρόβλημα αποθέματος και ένα πρόβλημα ροών. Υπάρχουν ακόμη αυλήρωτα ποσά από το 2013. Και το ίδιο πρόβλημα θα είναι ότι θα επανεληφθεί στο τέλος του 2014. Επ' αυτού λοιπόν έχουμε προβλεπόμενη συνάντηση στην ομάδα υψηλού επίπεδου για τους δημόσιους λογαριασμούς. Θα συναντηθούμε στις 24 Σεπτεμβρίου με τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συζητήσουμε αυτή την κατάσταση. Αλλά αν δώσω πίστη σε κάποια από τα σχόλια που έχουν ακουστεί, τα πράγματα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα. Κάποια κράτη ε, αποστέλουν αρκετά καθυστερημένα τους λογαριασμούς. Κάποιοι αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ε, αλλάζοντας τις ημερομηνίες τον Εύρο και τον Δεκέμβριο ώστε να προλάβουν το δημοσιονομικό έτος, αλλά έτσι δεν γίνεται ε, να καλυφθούν ε, οι πληρωμές με 60 μέρες διαφορά μεταξύ της στιγμής πληρωμής και της άφηξης των λογαριασμών. Χρειάζονται λοιπόν ε, περαιτέρω διερευνήσεις για να είμαστε βέβαιοι για το τι λέμε. Και θα πρέπει να μας τα πούν αυτά με περισσότερα στοιχεία και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι πρόσωποι των κρατών για να έχουμε μια σαφή εικόνα του τι γίνεται με τα απλήρωτα ποσά. Διότι μπορεί να λέμε τελικά εύκολα κάποιες φορές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα βρεθεί μια λύση, αλλά φαίνεται τελικά να ε, τραβάμε ένα σκηνή που κάποια στιγμή θα το σπάσουμε. Αυτά ως προς το αποθεματικό μας, ε, ως προς τις ροές. Δεν ξέρω αν είναι ε, σωστό αυτό που λέω, ίσως να είμαι αφελής ως νέος βουλευτής εδώ, αλλά στο μέλλον φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα απόσταση μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών που θα διονύζεται. Ίσως λοιπόν μια ιδέα είναι, και δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό, αλλά ίσως θα πρέπει να μειώσουμε τις υποχρεώσεις και ως προς τις προτεραιότητε, ε, θα δείξω εμπιστοσύνη προς τις διάφορες πολιτικές ομάδες ώστε να τις ιεραρχήσουμε καλύτερα στην ε, συνάντησή μας στις 29-30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου θα εξετάσουμε τις σχετικές τροπολογίες που όπως και εσύ, εσείς μας είπατε κυρία εισηγήτρια είναι πολλοί αριθμές αλλά θα πρέπει να τις δούμε κατά λεπτός. Τώρα για πριν περάσουμε στη συζήτηση που ήθελα να σας προτείνω και για τους ερχόμενους μήνες, το λεγόμενο brainstorming για τα θέματα του προπολογισμού, να δούμε και τις επόλοιπες εκθέσεις για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην Πατρίσια Σουλίν, η οποία θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσης για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την ε, περιοχή της ε, κοινότητας της Βαλένθια με κινητοποίηση ενός εκατομμυρίου 19.184 ευρώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν παραμείνει στην αίθουσα. Ε, χρειάστηκαν πληρωμές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να ε, επανενταχθούν όσοι απολύθηκαν από την μεταλλουργία της ε, περιοχής Κομμουνιτάς Κομινοτάδη-Βαλεντιάνα και το ποσό είναι 1.019.184 ευρώ. Επλήγει ε, σοβαρά η περιοχή ε, και είχε υποβληθεί και νωρίτερα έτοιμα στο Ταμείο. Από το Δεκέμβριο 2013 απολύθηκαν από 142 επιχειρήσεις 633 ε, άνθρωποι στη συνέχεια Ανάμεσα στο 2008 και 2012 χάθηκαν περίπου 15.000 θέσεις απασχόλησης. Ε, το πλεονάζον προσωπικό ε, στη μεταλλουργία προέκυψε από την οικονομική κρίση τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Προσαρμογής ε, ε, στην Παγκοσμιοποίηση στοχεύουν στην κάλυψη 300 απολυμένων. Πρόκειται για προσωπική βοήθεια προς πλεονάζοντες ε, με τη μορφή κατάρτισης, πρόθεσης του επιχειρηματικού πνεύματος και ούτω καθεξής. Οι ισπανικέ Αρχές άρχισαν τον Ιούνιο του 2014 να εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα για να ε, παρασχεθεί γρήγορα ε, βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. που για το 10ο αίτημα για το 2014, το Μάρτιο του 2015 υπέβαλε το αίτημά της η Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τον Αύγουστο του 2012 εξέδωσε τη γνωμοδότησή της και χρησιμοποίησε τα κριτήρια του κανονισμού για τη λειτουργία ε, του Ταμείου ε, Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Εμεί συμφωνούμε για τη χορήγηση βοήθεια ε, προ την Ισπανία επί τη βάση αυτού του κανονισμού. Επίση, θα ήθελα να λάβω σχόλια και παρατηρήσει από πλευρά σα και θα καταβάλω καθημερινή προσπάθεια για να τα ενσωματώσω στην τελική μου γνωμοδότηση. Πρόεδρο ευχαριστούμε την εισηγήτρια για τις διευκρίνήσει Υπάρχουν παρατηρήσεις, υπάρχουν σχόλια. Όχι. Θα εξετάσει η Επιτροπή της Τροπολογίας, αν υπάρξουν, και ε, στις 6 Οκτωβρίου ψηφίζουμε. 6-7. Ο Πολ Ρούμπι θα έρθει τώρα που θα μας παρουσιάσει ε, την ε, πρόταση για ε, την Γάνδη στο Βέλγιο. Α, ο κύριος Φερνάντες θα μας την παρουσιάσει. Δεν είναι εδώ ο κύριος Ρούμπικ. Πρόκειται για μια έκθεση που προβλέπει 570.945 ευρώ για το Βέλγιο στις 23 Δεκεμβρίου 2014 2013 13 ε, ε, μάλλον υπευλήθη αρχική ένταση και συμπληρώθηκε το 2014 ε, και η νομοθεσία Μάλλον η αίτηση ε, συνάδει με όλες τις νομοθετικές διατάξεις για τη λειτουργία του Ταμείου της ε, ε Παγκοσμιοποίησης ε, και προτείνουμε να εγκριθεί. 29 Σεπτεμβρίου ήταν, 29 Σεπτεμβρίου ήταν η ημερομηνία όπου ξέπνωσε η Πρόθεσμή για τις τροπολογίες και αναμένεται η έγκριση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών 6-7 Οκτωβρίου και στις 20 Οκτωβρίου θα περάσει το θέμα από την Ολομέλεια. Ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες. Υπάρχουν σχόλια. Παρατηρήσεις. Όχι. Ωραία. Τώρα θα μπορέσουμε να περάσουμε στο σεμινάριό μας, το λεγόμενο brainstorming. Θα γίνει και κλεισμένον των θυρών αυτή η συζήτηση. Κατά συνέπεια, όσες και όσοι δεν είναι συνεργάτες των μελών της Επιτροπής μας, θα παρακαλούσα να αποχωρήσουν. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας αυτή την αρχή του πρωινού της σημερινής ημέρας.